μια ανακοίνωση που αφορά τη νέα γαλλική κυβέρνηση. Μετά από τον διορισμό δύο εκ των συναδέλφων μας, ε, τη κυρία Σεσιλού Γκουλάρ ω Υπουργού ε, Ενόπλων Δυνάμεων και τη κυρία Μαριέλ Ντεσαρνέ ω Υπουργού υπεύθυνη ε, για τα ευρωπαϊκά ζητήματα στο Υπουργείο για την Ευρώπη και τις εξωτερικές υποθέσεις, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει την κένωση των θέσεών του, την εκένωση των θέσεών τους από τη 18η Μαΐου του 2017. Τους εύχομαι και στις δύο συγχαρητήρια και κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.